Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ εκεί πίσω στις φθηνές θέσεις, στα ορεινά. θα επιθυμούσα να κηρύξω την έναρξη της ακρόασης με την υποψήφια οριστής Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μογκερίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα ενώπιόν μας και χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και που είχαμε την ευκαιρία να Έχουμε και σε προηγούμενη ευκαιρία ως ε, εκπρόσωπος της Ιταλικής κυβέρνησης μας είχατε απευθύνει το λόγο. Θα ήθελα να θυμίσω ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου, αξιολογούμε τη γενική επάρκεια των υποψηφίων επιτρόπων, την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης αξιολογούμε τη γνώση σχετικά με το επικείμενο χαρτοφυλάκιο και τις επικοινωνιακές ε, ικανότητες. Έχετε λάβει ε, email τις γραπτές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που εν μέρει έχει συντάξει και η Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας θυμίσω πώς θα διεξαχθεί η ακρόαση αντίστοιχα με την ακρόαση με τον προτινόμενο Επίτροπο Χάν θα κληθεί η κυρία Μαγκερίνη να κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση που δεν θα ξεπεράσει τα 15 λεπτά και στο τέλος της συνεδρίας 5 με 10 λεπτά για να κλείσει θα έχει την ευκαιρία για δευτερολογία και 45 θα είναι ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Πρώτος γύρος από τους προσώπους των πολιτικών ομάδων και των μιαγεγραμμένων και στη συνέχεια οι πρόεδροι των Επιτροπών ΣΕΝΤΕ, ΙΝΤΑ και ΝΤΕΒΕ. Αυτά τα 11 μέλη θα έχουν ένα λεπτό για να κάνουν την ερώτηση και ε, μετά την απάντηση θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν και μια συμπληρωματική ερώτηση 30 λεπτό με ένα λεπτό απάντηση. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη, μία ερώτηση ενός λεπτού και μία απάντηση δύο λεπτών κάθε φορά. Οι πολιτικές ομάδες έχουν το χρόνο αγόρευσης και θα παρακαλούσα να σεβόμαστε όλοι το χρόνο μας, αλλιώς θα έχουμε δυσκολίες. Νομίζω στην ακρόαση με τον Επίτροπο Χάν τα πήγαμε καλά. Από τη φωνή μου ακούτε ότι απόψε έχω πρόβλημα να μιλήσω. Και επειδή δεν θα μπορώ ούτε καν να σας διακόπτω γιατί δεν βγαίνει η φωνή μου, απλώς θα σας κόβω το μικρόφωνο. Και παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας και επειδή έχω βραχνιάσει, παρακαλώ δείξε κατανόηση και μην λέτε τώρα τελειώνω, θα αρχίσει την τελευταία μου πρόταση γιατί θα σας κόβω νωρίτερα. Νομίζω ότι μπορούμε να τηρήσουμε το χρόνο μας όλοι κανονικά. Μετά τη συζήτηση, η οριστής επίτροπος θα έχει 5 με 10 λεπτά στη διάθεσή της για τα συμπεράσματα και να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση. Κυρία Μογκερίνη, μεγάλες προσδοκίες εναποθέτουμε στη θητεία σας. Έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία. Ήταν μια δοκιμαστική περίοδος, έτσι θα τη χαρακτήριζα, της πολιτικής των τριών ιδιωτήτων. Θέλαμε να έχουμε συνέργειες και είπα το εκπρόσωπος ταυτόχρονα είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Είναι πλήρης επίτροπος δηλαδή και ηγεσία ε, του συνόλου των επιτρόπων που ασχολούνται με τις εξωτερικές υποθέσεις και επίσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, που έχει λάβει ήδη μεγάλες διαστάσεις, να μπορεί να συντονίζεται με τις 140 αντιπροσωπείες στις διάφορες χώρες και να παράγει τόσο έργο ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα περιεχόμενο και να λαμβάνει υπόψη του τα τεκτενόμενα και τα αποφασιζόμενα και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Θυμίζω ότι εκεί χρειάζεται, απαιτείται ακόμα ομοφωνία και καλείστε να δείξετε ηγετική ε, στάση για να συγκεραστούν όλα τα συμφέροντα προς όφελος της ειρήνης ε, και της ελευθερίας παντού και στην άμεση γειτονία μας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες οι καιροί που έχετε την ευκαιρία να λάβετε μια τέτοια θέση. Θυμίζω ότι έχουμε μια σειρά ερωτήσεων και ζητημάτων που πρέπει να υλοποιηθούν σε ό,τι αφορά τα κοινοβουλευτικά δικαιώματα σε αυτό το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής. Ανέκαθεν ε, λέγαμε ότι η εξωτερική πολιτική είναι αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά το Κοινοβούλιο κάνει λόγο για κοινοβουλευτική δημοκρατία, για έλεγχο της πληροφορίας, έγκαιρη διαβούλευση, καθώς επίσης και ε, καλούμεθα να ακυρώσουμε και να επικυρώσουμε τις συνθήκες που συνάπτουμε και τις συμφωνίες και ε, αποφασίζουμε και για τον προπολογισμό. Λοιπόν, εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία και από τις συζητήσεις που είχαμε είμαι αισιόδοξο ότι θα καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα. Με χαρά λοιπόν Περιμένω τη συζήτηση. Επίσης γνωρίζετε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, στη στελέχωση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης όταν αποφασίσαμε τον κανόνα 1 τρίτο, 1 τρίτο, 1 τρίτο να μην είναι οι κεφαλές μόνο η ηγεσία ε, των κρατών μελών και το πεζικό για να το πω έτσι από ε, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και θα πρέπει κάποιος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει αποσταλεί να είναι στις ηγετικές θέσεις ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Νομίζω έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε, επαναλαμβάνω, με λογικό τρόπο και αποτελεσματικό, όσο και επικοδομητικό τη συνεργασία μας. Έχετε το λόγο κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, παρακαλώ.